Παρακαλώ καθίστε, κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση η οποία διακόπηκε στις 5 ε, Ιουλίου. τα πρακτικά της συνεδρίασης της 5ης Ιουλίου έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε